στην Επιτροπή όσον αφορά τον ρόλο τοπικών περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Τον ε, λόγο έχει η κυρία Μιχαήλοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Η νομοθεσία, η κείμενη, ζητεί από τα κρατημέλη να προβλέψουν ώστε να υπάρχουν κατάλληλε ε, προποθέσει. Και έτσι να υπάρχει διαβούλευση με τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, όπου υπάρχουν ε, εταιρικέ συμφωνίε και διάφορα λειτουργικά πηγαιρισιακά προβλήματα. Αυτέ οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ είναι πιο κοντά στον κόσμο και στον πολίτη, γνωρίζουν τι προβλήματα υπάρχουν και έχουν ένα πλεονέκτημα. Έτσι, μπορούν να διαμορφώσουν τι κατάλληλε πολιτικέ και έτσι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Επίση έχουν την αρμοδιότητα τη ε, απασχόληση. μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, ε, στι μεταφορέ κλπ. κλπ. Από την άλλη μεριά, αυτές οι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ δεν έχουν του απαραίτητου πόρου. Επομένω, χρειάζονται περισσότερη στήριξη από τον προπολογισμό περισσότερη συγχρηματοδότηση. Με την ε, υλοποίηση της πολιτικής συνοχής η διαβούλευση με τις αρχές αυτές έχει όλος μεταβληθεί διότι κάποια κράτη-μέλη δεν τηρούν αυτή την αρχή της εταιρικής σχέσης, της συνεργασίας ακριβώς όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία και στα κράτη που έχουν ομόσπονδιακή δομή δεν υπάρχει αυτή η κατάλληλη ισορροπία, δεν έχουν λέγει για τις πολιτικές αυτές. Οπότε θα πρέπει να αναβαθμιστεί η δυνατότητα αυτών των αρχών. Αυτό είναι το κλειδί για να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός αλλά και καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων. Και ισχύει επίσης για την πολιτική των ε, διαρθρωτικών και των ταμείων συνοχής. Επομένως, ε, αυτό αφορά και τις νεοφύς ε, επιχειρήσεις. Υπάρχει στρατηγική για την εξειδίκευση και όλα αυτά είναι καινούργιες πολιτικές. Αφορούν και την καινοτομία. Όλα αυτά είναι θετικά. Έχουμε την δήλωση του 15 Εγκρίθηκε από το άτυπο Συμβούλιο Ανάπτυξης. Ε, πρόκειτο επίσης για, για την δήλωση της ε, ε που στη συνέχεια οδήγησε στην συμφωνία του Άμστερνταμ που θα πρέπει όμως να υλοποιηθεί με συγκεκριμένες στρατηγικές για τις πόλεις. Τελευταίο αλλά σημαντικό, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν να σημαντικό ρόλο όσον αφορά κάποια συνεργασία διασυνοριακή, κάποιες πρωτοβουλίες που υλοποιούν την συνεργασία. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στα ερωτήματα του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της ε, Περιφερειακής Επιτροπής. Δηλαδή συγκεκριμένα τι θα κάνετε για να βοηθήσετε αυτές τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ούτως ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους ούτως ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν θετικά την διαχείριση ε, αυτών των ε, ταμείων, των διαφορετικών και επενδυτικών για την περίοδο 14-20. Θα πρέπει φυσικά να σεβαστούμε τις αρμοδιότητες αυτών των αρχών αλλά και τις ιδιωτυπίες του κάθε κράτους μέλους και έτσι να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη και βιώσιμη απασχόληση. Δεύτερον, για πέστε μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ξεκινήσει μια δημόσια πλατιά διαβούλευση κατόπιν ε, του, του, του, θέματος που επισημάνθηκε για την αναβάθμιση των τοπικών και περιφερειακών αργών. Έχουμε αυτά τα δύο ερωτήματα. Επίσης σας τονίζω ότι για την Επιτροπή Βεβαρικής Πολιτικής αυτά τα ζητήματα, αυτέ οι ερωτήσει είναι πολύ σημαντικέ. Γιατί θεωρούμε ότι ε, τοπικέ περιφερειακέ αρχέ είναι το κλειδί για την επιτυχία τη ε, Επιτροπή, συγγνώμη, τη πολιτική συνοχή. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε απασχόληση και ανάπτυξη. Τοπικέ και αρχέ ε, Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τον προγραμματισμό τη Επιτροπής ε, τη πολιτική συνοχή μετά το 2020. Περιμένω να μου απαντήσετε κύριε Επίτροπε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κυρία Μιχαήλοβα για τώρα. Τον λόγο έχει η κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Μιχαήλοβα, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω σε αυτή την προφορική ερώτηση εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικεντρώνεται στο ρόλο των ε, περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ε, διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ΕΔΕΤ. Γνωρίζετε ποια είναι η δική μας άποψη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ε, για να συνεργαζόμαστε αγαστά με τη ΣΟΤΑ και τις περιφερειακές αρχές που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία αυτά. Τα προγράμματα αυτά φέρνουν πιο κοντά τις περιφέρειες και τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα πρέπει να πιάνουν τόπο και να χρησιμοποιούνται με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποντάρει πάρα πολύ ε, στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση επιτόπου. Ξέρουν τι χρειάζονται οι περιφέρειες, ξέρουν τι μπορεί να γίνει, ξέρουν τι δεν μπορεί να γίνει. Η περιφερειακή πολιτική έχει αυτό το βασικό και θεμελιώδες χαρακτηριστικό. Υπηρετεί τις ε, ανάγκες του κάθε τόπου. Με τη δική σας υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, καταφέραμε να πείσουμε τελικά τα κράτη-μέλη να ε, εμπλακούν και οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές στην ίδια τη λήψη των αποφάσεων και σε προνομοθετικό στάδιο και καθ' όλη τη ε, διάρκεια της προγραμματικής περίοδου. Ε, χαίρομαι γι' αυτό και ε, ευγνωμονώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με το νέο τώρα κανονισμό έχουμε προαπαιτούμενο τη σχέση, τη, αυτή την εταιρική, τη συμμετοχή των αρχών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Δεν θα πρέπει να αποφασίζει μόνο η κεντρική κυβέρνηση. Αυτό τώρα πια έχει κατακτηθεί. Η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Υπάρχουν χώρες με παράδοση τέτοια συνεργασίας με τις περιφερειακές αρχές και άλλες χώρες που δεν το έχουν ακόμα τελείως καταλάβει ούτε ενσωματώσει την πολιτική τους. Χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό και όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις που έγιναν για τα ΕΣΠΑ και τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης αλλά και την υλοποίηση των έργων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό τον καιρό ε, κάνει μια μελέτη για να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτή η εταιρική σχέση και η πολυεπίπεδη λεγόμενη διακυβέρνηση κατά την ε, προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σας διαβεβαιώ ότι θα σας διαβιβάσουμε τους επόμενους μήνες τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Σε ό,τι αφορά τις ολοκληρωμένες ε, αστικές δράσεις, αναφερθήκατε σε αυτές κυρία Μιχαήλοβα και είναι και πάρα πολύ σημαντικές για την περίοδο 2014-2020 15 δισεκατομμύρια έχουν δεσμευτεί για τις αστικές περιοχές και τη δική τους ανάπτυξη. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί με τρόπο άμεσο της πόλης. Αυτή είναι μια απόφαση που δείχνει ότι εμπιστευόμαστε τις πόλεις, μπορούν οι δήμοι να ε, αποφασίζουν ποιες είναι οι ανάγκες τους και να δαπανούν αυτά τα κονδύλια. Τα ίδια ισχύουν και για τις δράσεις ε, της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και εκεί ε, καλείται ο δημόσιος τομέας να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό και την κοινωνία των πολιτών. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου έτσι ώστε η ατζέντα για τις πόλεις να υλοποιηθεί και να έχουν πραγματικό λόγο και οι Δήμοι και να συνομιλούν άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί η φτώχεια στις πόλεις ή να ε, βελτιωθεί η ένταξη των μεταναστών. Κυρία Πρόεδρε, εσείς αναφερθήκατε στην ε, ε, διακήρυξη, στην ανακοίνωση της Ρήγας. Υπάρχει και η δήλωση το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Όπως είπα, βοηθάει πάρα πολύ. Η Ολλανδική Προεδρία έχει εστιάσει στην αστική ανάπτυξη στο Άμστερνταμ το Μάρτιο έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση των ε, Δήμων που θα ε, καταλήξει στη διακήρυξη του Άμστερνταμ. Ε, συμφωνούν όλοι ότι χρειάζεται ένα αστικό θεματολόγιο, μια ατζέντα για τις πόλεις δηλαδή. Μέχρι τώρα οι χώρες επικαλούνται την αρχή της επικουρικότητας και δεν ήθελαν ευρωπαϊκό πλαίσιο ειδικό για τις πόλεις και την αστική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προτίθεμαι να διοργανώσω συνεδρίαση με δημάρχους ε, αρχής γενομένης από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν τα περισσότερα προβλήματα ε, με το προσφυγικό τώρα. Πέρα από την εκάστοτε εθνική πολιτική για την υποδοχή των προσφύγων, υπάρχουν δήμαρχοι που καλούνται να λάβουν έκτακτα και πήγοντα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και τις ε, νέες προκλήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τις πόλεις αυτές, οι οποίες πλήττονται περισσότερο και έχουν τα οξύτερα προβλήματα, λόγω της μαζικής άφηξης προσφύγων. Βοηθούμε λοιπόν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να αξιοποιήσουν όσο μπορούν ε, και στο μέγιστο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Συμφωνείτε φαντάζομαι μαζί μου ότι το χρήμα δεν είναι το παν. Δεν αρκούν τα κονδύλια. Χρειάζεται διοικητική ε, δυνατότητα, ικανότητα απορρόφησης, τα έργα να πετυχαίνουν, να γίνονται τα σωστά έργα. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς από τις Βρυξέλλες τι πρέπει να γίνει στην περιφέρεια. Αυτό είναι πάρα πολύ αποφασιστική σημασία και η χρονιά αυτή, το 2016, είναι επίσης αποφασιστική. Χρειάζονται ε, βιώσιμα έργα που να απαντούν πραγματικά στις ανάγκες των πολιτών. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ε, προβλέψεις για να ενισχύονται οι δυνατότητες απορρόφησης και ε, μάλιστα 5 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2014-2020 και είμαι βέβαια ότι θα βοηθήσει αυτό και την οικονομική κατάσταση και θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπη. και τώρα έχουμε δει πανηγάσεις από πλευράς των πολιτικών ομάδων και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τον λόγο ο κύριος Φανίστρη Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Κρατή. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, για τόσα είπατε δηλαδή. Όντως, τρία σημεία θέλω να θίξω. Πρώτον, για τις περιφέρειες. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει τάση επαναθνικοποίησης, διαπιστώνουμε. Δεύτερον, η αρχή της εταιρικής σχέσης, άρθρο 5 του κανονισμού, δεν εφαρμόζεται πλήρως όλες τις χώρες. Εξακολουθούν κάποιες περιφέρειες να μην έχουν ισότιμη αντιμετώπιση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τρίτον, η Επιτροπή των Περιφερειών ρητά ανηφέρει την ε, κεντρική διάσταση, την ε, τάση δηλαδή της κεντρικής διαχείρισης. Το ΕΛΚ λοιπόν ζητάει η επικουρικότητα να τηρείται πλήρως. Και το ε, ερώτημα είναι, είπατε, αναφερθήκατε στη μελέτη, θέλουμε και εμείς με το άρθρο 6.3 να δουλέψουμε βάσει αυτού και θέλουμε σε αυτό το θέμα να μπούμε περισσότερο σε βάθος. Λοιπόν, επ' αυτού μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο θα ζητήσετε μια δημόσια διβούλευση για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici. Για τη σοσιαλιστική ομάδα. Το λόγο έχει η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πίτρο, συνάδελφοι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό να γίνεται αυτή η συζήτηση και είναι πάρα πολύ εύστοχο και αυτό το ψήμα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που για άλλη μια φορά επιβεβαιώσατε το, τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, ε, ιδίως όσον αφορά την διαχείριση της πολιτικής συνοχής από πλευράς των πόλεων. Γνωρίζουμε ότι η πολιτική της συνοχής σήμερα είναι το βασικό εργαλείο για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το πρόγραμμα Juncker. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο. Την δε επόμενη περίοδο προγραμματισμού που έχουμε αρχίζει και θα τη συζητήσουμε σύντομα. Είναι κάτι που θα πρέπει να κρυθεί και να διασκεδαστούν οι ανησυχίε που υπάρχουν διότι εάν δεν έχουμε κάποιο είδου αλλαγή του προγραμματισμού και η περικοδότηση δεν αυξηθεί, τότε πρόκειται να έχουμε συρρήγνωση των πόρων για, τους, για τις κατηγορίες αυτές που ακριβώς χρειάζονται αυτοί οι πόροι. Θα πρέπει ε, να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα όλες οι πόλεις. Ε, οπότε θα πρέπει οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ε, θα πρέπει να εμπλακούν μέχρι το τέλος του περίοδου προγραμματισμού. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια στην πολιτική των Ευρωπαϊκών Ταμείων και θα πρέπει η πολιτική της συνοχής να συνεχίσει να είναι η ατμομηχανή για ανάπτυξη και απασχόληση. Ακριβώς όπως να το σήμερα, οπότε γι' αυτό σας παρακαλούμε εσείς να είσαστε ο σημειοφόρος για αυτή την υπόθεση των τοπικών και περιφερειών αρχών. Για το ΙΣΙΑ έχει το λόγο ο κύριος Πιοτρόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, ως στόχο μεταξύ άλλων και τη βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη. Θα πρέπει να μειωθεί η ψαλίδα ε, που υπάρχει μεταξύ των πιο φτωχών και των πιο πλούσιων περιφερειών. Πολλές φορές υπάρχουν κονδύλια, αλλά δεν μπορούν να τα απορροφήσουν οι αρχές της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το πρόβλημα δεν είναι η συγχρηματοδότηση, η συνυπευθυνότητα, ε, ε, αλλά ε, η προστιθέμενη αξία 2014-2020. Ε, Πολλές φορές οι περιφέρειες ε, και οι τοπικές αρχές δεν ξέρουν ε, πώς να υποβάλουν την αίτηση για να πάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η συγχρηματοδότηση, είναι η προστιθέμενη αξία. Εγώ προέρχομαι από την Πολωνία και στη δική μου περιφέρεια οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ζητούν λύση και με περισσότερη ευελιξία στη χρήση των κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη από τις εταιρείες. Αυτό θα δώσει όθηση για περισσότερη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και επενδύσει Γιάκοφτσι από τους φιλελευθέρου. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρέπει να πω καταρχάς ότι ε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Μιχαήλοβα και τους άλλους συναδέλφους ε, από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες που προώθησαν αυτή την υπόθεση. Εγώ έχω στήσει όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία στην ενίσχυση ε, των πόλεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαρχιών. Για μένα αυτό ε, σήμαινε υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους. Τώρα θέλω να τονίσω ότι... Είμαι ακράδαντα πεπισμένο ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση προς την αρχή της επικουρικότητας πρέπει να γίνει σεβαστή. Γνωρίζουμε ποια είναι η ευρωπαϊκή πρακτική. Όσο πιο αποκεντρωμένες είναι οι χώρες, όπως η Δανία Φερρυπίν, ε, τόσο το καλύτερο. Ε, έχουν την υψηλότερη ανάπτυξη και το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Όσο πιο συγκεντρωτική είναι μια χώρα, όπως η Κροατία ή η Ελλάδα Φερρυπίν, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα της ανάπτυξης. Εμείς χρειαζόμαστε ε, να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και για την απορροφητικότητα. Έχουμε μια κατάσταση όπου χώρες υπερβολικά συγκεντρωτικές δεν ε, είναι σε θέση να απορροφήσουν τα υφιστάμενα κονδύλια. Αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Γι' αυτό οι πόλεις και οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε να έχουν και ανταγωνισμό μεταξύ τους, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, με τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Αν υπήρχε άμεση πρόσβαση των πόλεων και των ε, ΟΤΑ θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. και θα αυξανόταν και η ποιότητα ζωής πολλών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλές πόλεις και περιφέρειες. Θέλω να προσθέσω και μια άλλη ανάγκη που υπάρχει, διεθνούς συνεργασίας, διασυνοριακής, το Ιόνιο και η Αδριατική είναι εξαιρετική η δική μου περιφέρεια. Και τέλος ε, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να προχωρήσει το θέμα χάρη σε αυτή την προφορική Από την ΚΟΕ το λόγο τώρα έχει ο κύριος Παπαδημόλης Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, χρειάζεται η κυρία Κρέτσου όντως μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων. Μεγαλύτερη αποκέντρωση. Λιγότερο συγκεντρωτισμός. Λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερο μερίδιο από την από τα διαρθρωτικά ταμεία και από τα σχετικά κονδύλια για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αλλά κυρίως χρειάζεται και μεγαλύτερη βοήθεια και τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν σε διάλογο με τις εθνικές αρχές στις τοπικές και περιφερειακές αρχές γιατί πολύ μικροί δήμοι ή περιφέρειες δεν έχουν την τεχνογνωσία και τη διοικητική επάρκεια να καταθέσουν προτάσεις να καταθέσουν φακέλους και φυσικά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα και σε χρήματα και σε τεχνική βοήθεια για εκείνες τις πόλεις τα νησιά τις περιφέρειες που δίπλα στα μόνιμα προβλήματά τους αντιμετωπίζουν και την όξυνση της κρίσης του προσφυγικού. στην ελλάδα έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην πρωτεύουσα της χώρας την αθήνα. περιμένω λοιπόν με ενδιαφέρον και τη διαβούλευση και τις προτάσεις της ε, κομισιόν γιατί πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος στην πράξη και με τεχνική βοήθεια και με χρήματα οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην αξιοποίηση των τοπικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. από τους Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα αυτό, επίκαιρη ερώτηση σε καιρούς οικονομικής κρίσης, προβλημάτων ανάπτυξης και ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα αν δεν χρησιμοποιούσαμε το δυναμικό και των περιφερειακών περιοχών και των ε, τοπικών αρχών. Η δομή βέβαια των χωρών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Όμως σε πολλές περιπτώσεις η ανταλλαγή βέλτιστων ε, πρακτικών πρέπει να θαρρύνεται. Ζητάω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει αυτή την πρακτική ανταλλαγής βέλτιστων ε, πρακτικών Επιπλέον, θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια μεθοδολογία για να αξιολογήσει την επάρκεια του διοικητικού μηχανισμού των χωρών μελών. Θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην ποιότητα της συμμετοχής των ε, τοπικών, αρχών στις αποφάσεις των χωρών και την επάρκεια των ιδίων πόρων και τη εντολής που έχουν οι τοπικές αρχές προκειμένου να εφαρμόσουν την περιφερειακή πολιτική. Οι εθνικές αποφάσεις στην περιφερειακή διάσταση πρέπει να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες. Η εταιρική σχέση επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει πραγματικά εταιρική σχέση ανάμεσα στην ε, κεντρική διοίκηση και τις τοπικές αρχές πολύ συχνά. Συχνά πρόκειται για κάτι καθαρά τυπικό που υπάρχει θεωρητικά, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται πιο κοντά στον κόσμο και μπορούν καλύτερα να εντοπίσουν τις ανάγκες και τα μέσα που χρειάζονται. Πολύ σημαντικό μάλιστα, δεδομένων και των διαφορών που υπάρχουν ε, από περιφέρεια σε περιφέρεια, εξαιτία μεταξύ άλλων των κλιματικών αλλαγών και του προσφυγικού. Ευχαριστούμε, ο κύριο Σταμάτο, έχει τώρα το λόγο. Η ε, κυρία Ταμάτο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική τη ε, συνογή για να πετύχει θα πρέπει να βασίζεται στην συνένεση και να υπάρχει συνεργασία σε κάθε επίπεδο μεταξύ δηλαδή περιφερειών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, ε, η σημερινή πολιτική να υπόψη ότι δεν λειτουργεί, γιατί θα πρέπει κάπω να γίνει και να μειωθεί η απόσταση μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διακυβέρνηση. Δεν υπάρχουν απαραίτητε διοικητικέ ικανότητε ε, για τη διαχείριση ε, ε, έχουν σωρευτεί πάρα πολλά αχρίαστα έργα και προγράμματα και επομένω το ίδιο και για την πατρίδα μου θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο στην πολιτική συνοχή οι περιφέρειε. Ε, Επίση, πέραν τη ανάλυση και του προγραμματισμού, θα πρέπει να προβληματιστούμε στο πώ θα γίνει ε, να αυξηθεί η απορρόφηση. Τελευταίος μήνες τα πράγματα είναι απίστευτα, οπότε επομένως θα, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια προγράμματα και να αυξηθούν οι πόροι και θα πρέπει να δούμε πώς θα εγκριθούν κάποια προβλήματα λειτουργικά και αυτά να καλυφθούν από την καινούργιο προγραμματισμό. Άρα θα πρέπει να εξομπιστούν καλύτερα οι περιφερειακές αρχές για αυτά τα προγράμματα και έργα, να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρώπη να συνδεθεί η πολιτική συνοχή με την οικονομική διακυβέρνηση για να καταπολεμηθούν τα ελλείμματα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα σημεία και νομίζω ότι υπάρχει συνένεση από όλες τις πολιτικές πτέρυγες. Ε, όμως θα πρέπει να δούμε τι κάνει η κυβέρνηση Ρέντζε. Ρέντζε διότι ε, ε, ασχολείται περισσότερο με την προκλογική εκστρατεία και οδηγόμαστε σε κάποιο είδου ε, πολιτική λιτότητα. Χρειάζεται μια πιο εύστοχη πολιτική συνοχή τώρα από την, ε, την Ομάδα Εθνών και Ελευθερίας. Ο κύριος Στούγκερ, ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σας. Πρόεδρε, σε δύο μήνες έχουμε δημοψήφισμα στην Ολλανδία για τη συμφωνία με την Ουκρανία και την περασμένη εβδομάδα φαίνεται ότι ο κύριος Σόρος, μέγας Αμερικανός επενδυτής, έχει στείλει 200.000 ευρώ για να χρηματοδοτήσει το στρατόπεδο του ΝΕ. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χοντρά οικονομικά συμφέροντα και υποστηρίζουν το ΝΕ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το δημοψήφισμα αυτό χειραγωγείται. Και από ό,τι φαίνεται η Ολλανδία είναι επανάπτυκτη χώρα ω προς τον εκδημοκρατισμό. Μια επανάπτυκτη χώρα, ε, και μιλάμε για περιφέρειες, ε, μια περιφέρεια είναι και η Ολλανδία, μπορούν να ε, έχουν κονδύλια από το Αναπτυξιακό Ταμείο. Και θέλω να σας ζητήσω κυρία Πρόεδρε να σώσετε τη δημοκρατία και να στείλετε αυτά τα λεφτά στο Ταμείο τη Εξαρτία του Όχι. Κύριε Στούγκερ, έχετε δύο μπλε κάρτε τώρα εσείς. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, λέει ο κύριος. Ο κύριο Βανίστερ Ρόι και μετά ο κύριος Έθριτ. Πολύ σύντομο θα είμαι. Ε, είμαι έξαλλος από την τοποθέτηση αυτή. Είναι η πανάπτυκτη περιοχή από πλευράς δημοκρατίας η Ολλανδία. Πώς μπορεί να εκπροσωπεί πολίτες Ολλανδούς και να καταχράτε αυτή την ημερήσια διάταξη. Εδώ συζητάμε περιφερειακή πολιτική και περιφέρειες. Κάτι πάει στραβά εδώ. Μπορείτε να μου απαντήσετε τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Έθριτς, για να απαντήσετε και στους δύο καλύτερα στη συνέχεια. Πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Έθριτς και να απαντήσετε και στους δύο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που δέχεστε και την ερώτηση κύριε Στόγκερ. Μιλήσατε για το δημοψήφισμα στις κάτω χώρες και τους μεγάλους επενδυτές και τις business που υποστηρίζουν την πλευρά του ναι. Ο κόσμος στην Ολλανδία θα το εκλάβει το δημοψήφισμα ως δημοψήφισμα υπέρ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε ότι έχουμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο δημοψήφισμα. Έχετε κανένα μήνυμα για το λαό του Ηνωμένου Βασιλείου. ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, τη στιγμή που μεγάλοι Αμερικανοί επενδυτέ, το λέω στον κύριο Βανίστερόι, μπαίνουν στον κόπο να ασχοληθούν με ένα δημοψήφισμα στι κάτω χώρε, χωρίς να κάνει τίποτα ελλανδική κυβέρνηση, ε, μπορούμε να πούμε ότι δημοκρατικά υπάρχει έλλειμμα εκεί. Γιατί περί αυτού πρόκειται και το ανέφερα ακριβώς αυτό το δημοψήφισμα. Και καλό είναι λοιπόν να προσέχουμε ε, τα που ακούμε. Και απαντώ στον κύριο Έφριτς τώρα, Βεβαίως, ο Ολλανδικός λαός βλέπει το δημοψήφισμα αυτό ως ευκαιρία για να βγάλει όλα του τα αποθυμένα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα στρεβλά που συμβαίνουν. Και ελπίζω να είναι συντριπτικό το όχι και καλό το αποτέλεσμα. Και αυτό θα είναι ένα προήμιο, αν θέλετε, για τα όσα θα ακολουθήσουν ε, στη συνέχεια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος οι τοπικές και περιφερειακέ αρχέ στη σημερινή ευρώπη αποτελούν ίσω το βασικό κύτταρο πάνω στο οποίο θα πρέπει να επανοικοδομήσουμε τα κράτη τη Ευρώπη. οι αρχέ αυτέ σε χώρε όπω η ελλάδα έχουν αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό όχι τόσο λόγω έλλειψη αρμοδιοτήτων αλλά κυρίω λόγω έλλειψη ανθρώπων. ο πληθυσμό έχει συρρυκνωθεί δραματικά με αποτέλεσμα τη σημερινή άσχημη κατάσταση. συμφωνώ λοιπόν απολύτω πω πρέπει να ενισχύσουμε την περιφέρεια και κυρίω του ανθρώπου τη, του αγρότε, του κτηνοτρόφου, όλους εκείνους που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην επαρχία. σκοπός μας πρέπει να είναι η αποκέντρωση με την οποία θα βελτιωθεί επίσης και η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα. δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση στην ελλάδα έχει βάλει στο στόχαστρο για να εξολοθρεύσει μεταξύ των άλλων κοινωνικών ομάδων και τους αγρότες. με την πολιτική της καθιστά λόγια άνευ περιεχομένου τα όσα συζητάμε σήμερα εδώ καθώς δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια αγρότες για να τους ενισχύσουμε. τέλος θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως όλοι οι πόροι χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων που θα διατεθούν θα πρέπει να διατεθούν με απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο μακριά από οποιαδήποτε υπόνοια διαφθοράς αν θέλουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα προς την ελλάδα στην οποία σήμερα υπάρχει πανελλαδική πανεργατική απεργία απέναντι σε μια μνημονιακή κυβέρνηση της αριστεράς η οποία συνεχίζει τα μνημόνια και εξαθλειώνει τις ζωές των Ελλήνων. Ευχαριστώ. Κύριε Τσέλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ξέρουμε ότι οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως στρατηγική του 2020 η ΟΤΑ και οι περιφερειακές αρχές ε, φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη ε, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα που έχουν. Όπως τώρα είναι η υποδοχή και η ένταξη και η στέγαση και η περίθαλψη ε, των μεταναστών και των προσφύγων. Άρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί οι Δήμοι και οι κοινότητε και οι περιφέρειες να συμμετέχουν πολύ περισσότερο στι συμφωνίε εταιρική σχέση, στα ΕΣΠΑ και στα διάφορα έργα, στα διαρθρωτικά ταμεία. Τώρα ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι δεν γίνεται αυτό πλήρως, ούτε έχουμε πετύχει. Το 5% που πήγαινε στις πόλεις δεν φτάνουν σε όλες τις χώρες και δεν φτάνουν σε όλες τις πόλεις κυρίως που είναι οι αποδέκτες. Ε, άρα τώρα καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι μόνο μια κλίση, είναι και κλίση αφύπνισης ε, για να υλοποιούνται σωστά τα προγράμματα αυτά και να ενισχύονται περισσότερο οι δήμοι, οι κοινότητες και οι περιφέρειες. Γιατί εκεί είναι τα προβλήματα και εκεί μπορεί η ευρωπαϊκή πολιτική να πιάνει τόπο και η ευρωπαϊκή συνοχή να είναι ορατή. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια περώτηση για σας κύριε Τζέλερ. Θέλετε να απαντήσετε βεβαίως λέει. Κύριε Τζάνι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, συμφωνώ με την συμμετοχή των τοπικών αρχών στη διαχείριση των κονδυλίων αυτών, αλλά και άλλων. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Πώς μπορούμε να βγάλουμε τα πολιτικά κόμματα και την ανάμειξή τους σε αυτή τη διαδικασία και τελικά να επωφελούνται εκείνα από τα κονδύλια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Παρακαλώ για να απαντήσετε. Κοιτάξτε, και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές παίζει ρόλο η πολιτική. Αλλά το πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια που υπάρχουν στην περιφερειακή πολιτική, αυτό το λένε οι κανονισμοί. Είναι σαφές. Και υπάρχουν διατάξει και λογοδοτούν οι εκάστοτε αρχές. Εγώ δεν έχω ε, γνώση ότι υπήρξε κατάχρηση για κομματικούς σκοπούς τέτοιων κονδυλίων, αυτό θα ήταν απάτη και κανονικά θα πρέπει να διωχθεί αρμοδίως. Μανσκούρ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας δεν λειτουργεί. Τώρα είναι εντάξει. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι που βλέπω ότι η σημερινή συζήτηση ασχολείται με το ρόλο κλειδί των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Όντως, οι πόλεις είναι πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης, άρα και αστικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, το 2015, 40% της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στι πόλεις. Χρειάζεται μια πολιτική λοιπόν για τις πόλεις που να είναι αποτελεσματική. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στις ανησυχίε του κόσμου στην Ευρώπη που βλέπει ότι δημιουργήθηκε χάσμα στην ανάπτυξη ανάμεσα στις αστικές και τις ε, περιοχές της υπαίθρου. Ιδιαίτερα τις άκρος περιφερειακές περιοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν ένα σωρό μειονεκτήματα. Η πολιτική συνοχής λοιπόν πρέπει να διατηρήσει το αρχικό της πνεύμα που ήταν η δαφική αλληλεγγύη, κάτι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτή την αρχή. Η συμπληρωματικότητα επίσης ανάμεσα στις διάφορες περιοχές είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται εγκάρσια αντιμετώπιση που να καθοδηγείται από την αρχή της επικουρικότητας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χωρών μελών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα ο κύριο, ε, κύριος Μπενίτο Θηλουάγα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να έχουμε κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσουμε τους πολίτες την απασχόληση αλλά και την αλλαγή την κοινωνική έτσι ώστε να έχουμε μια πιο βιώσιμη κατάσταση για την κοινωνία μας. Χρειάζονται επενδύσεις λοιπόν που να καλύπτουν αυτούς τους δύο στόχους και να λάβουμε υπόψη μας ότι πράγματι είναι τοπικές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν καλύτερα να εντοπίσουν τις ανάγκες και που πρέπει να κατευθυνθούν οι προσπάθειές μας. Γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε για τις επενδύσεις με συμμετοχή όλων. Όμως, τα διευθυντικά ταμεία και το επενδυτικό ταμείο από κοινού δεν θα πρέπει να αφήνουν την πόρτα ανοιχτή σε περικοπές και να μην δίνονται χρήματα στις πόλεις σε βάρος της υπαίθρου. Διότι η χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική και για τις ΜΕΝ και για τις ΔΕ και κυρίως για εκείνες τις περιφέρειες που έχουν κάποια μειονεκτήματα οικονομικά ή φυσικά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Έτεριτς. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζω ότι είσαστε ένας άνθρωπος λογικός, οπότε αυτό που θέλω να, να τονίσω το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Οπότε ίσως ε, μπορείτε να βρείτε να φερθείτε με δικαιοσύνη προς την περιφέρεια μου. Πρώτα-πρώτα, ε, στα δυτικά Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου έχουμε εξωθηθεί να, να, έχουμε κάποιο είδου μεικτή διοίκηση και το επίκεντρο τη πολιτική του είναι να χρηματοδοτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά γίνονται εγκρυπτό και απαραβίστο. Επιλήψιμα, ο κόσμο δεν έχει λέγην. Οπότε έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση αμαυρώνεται και όλα αυτά γίνονται με τι περιφερειακέ και τοπικέ αρχές. Όμως υπάρχει κάποια ευκαιρία να μπορέσετε να επιδείξετε την καλή σα διάθεση, καλή πίστη εκεί στα West Midlands, εκεί που θέλουμε βοήθεια. Οπότε έτσι ε, εμείς ξέρετε ότι δίνουμε περισσότερα από όσα παίρνουμε, οπότε ε, ρίξτε μια ματιά συνεργασία εμένα γιατί χρειάζεται ε, χρηματοδότηση. Είναι και θέμα κουλτούρας, πολιτισμού και αυτό ο υπόδρομος που χρειάζεται κάποια ενίσχυση θα είναι κάτι το θετικό για όλο τον κόσμο και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπη Κύριε Έθεριτζ λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει μια περώτηση μπλε κάρτα για σας. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εσείς είστε ένας εκπρόσωπος του λαού που έχετε μεγάλη επαφή με τους ψηφοφόρους σας και σας ερωτώ ε, για να δω και τι γίνεται στις κάτω χώρες. Όταν πάτε στην εκλογή σας περιφέρεια, ποιο είναι το κλίμα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη δουλειά τους τα τελευταία χρόνια, που είναι μέχρι το λαιμό καταχρεωμένοι, πληρώνουν πολλούς φόρους, τι αίσθηση έχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Γνωρίζουν καν αυτόν τον όρο περιφερειακή ανάπτυξη. Μαθαίνετε, ακούτε πράγματα εσείς από τους ψηφοφόρους σας. Στα δυτικά Μίτλαντ ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης. Τι είναι αυτά η συνοχή και τα λοιπά για να είναι πιο εύκολη η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτό που αισθάνονται είναι ότι θέλουν να είναι πιο ελεύθεροι γιατί ε, ψήφισαν σε μεγάλο βαθμό το δικό μου κόμμα και συχνά το κάνουν, αυτό που αισθάνονται είναι ότι δεν τους βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι δυσκολίες και τα δεινά που αντιμετωπίζει με την ανεργία, με τους μισθούς που έχουν συγκληρωθεί, με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, κάνουν τους ανθρώπους να είναι πάρα πολύ πικραμένοι, αισθάνονται τεράστια πικρία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν αυτό να αλλάξει, να απελευθερωθούν. Ε, ο κύριος ε, Μπριουά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπε η Κορίνα Κρέτσου και έχω ε, κάπως ανησυχήσει και θορυβηθεί γιατί βρισκόμαστε σε μια καμπή. Μεταφέρονται, χωρούνται αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη γιατί αυτό που επιζητούν τώρα είναι οι περιφερειακές αρχές να ε, αντικαταστήσουν τα κράτη. Ε, το ομολόγησε κάπως η Κορίνα Κρέτσου που είπε για τη μετανάστευση θα πρέπει να βοηθήσουμε καμιά φορά τις πόλεις πολλές φορές απέναντι και αντίθετα με τη γνώμη των κρατών μελών. Άρα αντιστρέφουμε την αλληλεγγύη και την κυριαρχία μάλλον και αυτό είναι απαράδεκτο. Αύριο ποιο θα είναι ο πολιτικό ρόλο των κρατών μελών όταν θα διαφωνούν βαθύτατα με μια τοπική αρχή. Τι θα γίνει. Τώρα περνάμε στο ΚΑΤΣΔΙΑ. Είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο και φοβούμαι ότι δεν μπορούμε να τους δώσουμε. Ε, είναι πάρα πολύ Νόβακοφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φανίστε για το έργο, για το ψήφισμα το οποίο έχουμε και την κυρία βέβαια Μιχαήλοβα για την στήριξή της. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός διαχειρίζεται από τις χώρες μέλη οι αρχές όμως είναι εκείνες, οι τοπικές, οι οποίες εφαρμόζουν τοπικά προγράμματα. Πολλά από τα χρήματα, πολλά από τα κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται για τέτοια τοπικά προγράμματα. Δεν μπορούν να επενδύσουν λοιπόν οι τοπικές αρχές. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές αρχές από το Α μέχρι το μεγα, να αναπτύσσουν προγράμματα, να τα εφαρμόζουν, να τα διαχειρίζονται με έναν ευέλικτο τρόπο. Πολλές χώρες δεν μπορούν να εφαρμόσουν προγράμματα γιατί δεν έχουν χρήματα και γι' αυτό θα έπρεπε να βασιστούν σε μηχανισμούς της χώρας. Σας παρακαλώ να σέβεστε το κάτι το χρόνο σα αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Κύριο Κοτσολίνο. Μια παρατήρηση μόνο θα ήθελα να κάνω προ την Επίτροπο. Είπατε ότι προοδευτικά ενισχύουμε το ρόλο των τοπικών αρχών. Δήμοι, περιφέρειες και καμιά φορά μακροπεριφέρειες. Και τώρα με την αστική ατζέντα το θεματολόγιο. Ταυτόχρονα προχωράτε με την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ε, προγράμματα ρυθμιστικά και ε, τι γίνεται με την πολιτική συνοχή και την επικουρικότητα. Έχουμε περιορισμούς ε, και στους προπολογισμού. Ποια είναι λοιπόν η νέα μορφή και ο ρόλος της συνοχής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε ε, και να το παρακολουθήσετε με προσοχή για να μην έχουμε ε, συγκρούσεις στο μέλλον ε, και αντικρουόμενες πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών τους. Γι' αυτό και πρέπει να μπορούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των αντίστοιχων κονδυλίων. Φοβάμαι όμως ότι σε πολλές χώρες μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν έχουν ούτε την εμπειρία, ούτε τις ικανότητες να διαχειριστούν τέτοια προγράμματα. Στις μεγαλύτερες χώρες, στις πιο ανεπτυγμένες, όπου υπάρχει αποκέντρωση, οικοδομούνται τέτοιες ικανότητες εδώ και δεκαετίες. Οι χώρες αυτές είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ότι μικρότερες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες μέλη προς την αποκέντρωση και προς την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όταν πρόκειται για την οργάνωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Έτσι, οι σημαντικές αποφάσεις, σημαντικές για τον κόσμο, θα λαμβάνονται πιο κοντά σε αυτούς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, λέει κύριο Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Κάθε επένδυση τελικά θα καταλήξει σε ένα δήμο, σε μια πόλη και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και στηρίζω τις προτάσεις των συναδέρφων προκειμένου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουν άμεσα πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να υπάρχουν κανόνες δηλαδή βάσει των οποίων οι κεντρικές αρχές να δίνουν τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν στην χρήση των κολυδιών αυτών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση σε βάρος περιφερειών ή πόλεων. Κανέκλεισε επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την βελτίωση της εφαρμογής αυτού του μηχανισμού. Έτσι, η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι είναι τώρα. Ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι αγαπητοί Επίτροπε. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι οι βασικέ αρχές τη πολιτική αυτή είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και οι εταιρικέ σχέσεις. Δυστυχώς πολύ συχνά αυτά στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε τα ΕΣΠΑ ε, που έχουν εκπονηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ενώ ε, η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν συμμετέχει καθόλου στην χάραξή του. Ε, θα πρότεινα λοιπόν στο μέλλον όταν συζητούμε για την πολιτική συνοχή να βάλουμε ένα κανόνα και ο κανόνας να είναι ότι για τα ΕΣΠΑ χρειάζεται περιφερειακή ε, απόφαση, να είναι των περιφερειών. Και οι περιφέρειες να έχουν και την ευθύνη της υλοποίησης, να είναι δική τους δουλειά. Είναι σημαντικό οι περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν από την αρχή στη ε, χάραξη των πολιτικών το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο επίσης να συνδυαστεί με την πολιτική συνοχής. Αλλά ερήμην των ΟΤΑ αυτά δεν γίνονται. Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι χρειάζεται να γίνεται αυτή η διαφούλευση και οι διαπραγματεύσει με τι τοπικέ αρχέ για τα λειτουργικά σε προβλήματα. Και αυτό όμω είναι κάτι το οποίο με τον χρόνο δεν βελτιώνεται. Γιατί μόνο το 1 τρίτο το 2015 το, το έκανε αυτό και τότε, μόνο, μόνο αυτό το τόν τρίτον μπόρεσε να καθορίσει τη συνεργασία με τι αρχέ, τη προτεραιότητας. όμω θα πρέπει να δούμε πώ θα υπάρξει ένα τέτοιο ε, πλαίσιο τόσο ώστε να γίνουν κάποιε επενδύσει ε, όπου χρειάζεται. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό οι τοπικέ και οι περιφερειακές να εμπλακούν σε αυτή τη φάση στην συζήτηση, διαβούλευση και παρακολούθηση και φυσικά υλοποίηση των προγραμμάτων. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα εμπλακούν όλοι οι οι εταίρε κοινωνία των πολιτών σε κάθε επίπεδο. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια τέτοια διαβούλευση για να αναβαθμιστεί ο ρόλο αυτών των αρχών και μετά επί αυτή τη βάση να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Επομένω, το κράτο μέλο θα πρέπει να συνεργαστεί με αυτέ τι αρχέ για να οδηγηθούμε σε απασχόληση, βιώσιμη αλλά και ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ, Χέντμαν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπα, κυρίες και κύριοι, τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν την αρμοδιότητα το 70% των ε, επενδύσεων του δημοσίου. Οπότε θα πρέπει να τους ε, αναγνωριστεί ο ρόλος για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, όμως θα πρέπει να τους δώσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ε, να μην είναι μόνο αυτοί που τυπικά εγκρίνουν και προσυμπογράφουν να έχουν ουσιαστικό ρόλο να αναγνωρίσουν επομένω την εμπειρία, τη γνώση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Μιλούμε τώρα για αυτό το ε, ταμείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις ε, τοπικές αρχές να βοηθήσουν στην ε, διαχείριση θα πρέπει να υπάρξει πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ περιφέρειας, τοπικού επέδου και Ευρώπης. Αυτό μόνο να ωφελήσει μπορεί την οικονομία. Τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε, ε, συνάδελφοι, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος, παρά το ότι πολλοί ακόμα έχετε ζητήσει το λόγο. Και τώρα δώσουμε τη σκητάλη στην κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή. Όσον αφορά εμένα, το ξέρετε ότι θεωρώ πως ο κύριος εταίρος μας όταν πρόκειται για την περιφερειακή πολιτική είναι πράγματι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οι πρόεδροι πάνω από 280 περιφέρειες βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση μαζί μας. Πράγματι είναι αυτοί που είναι πιο κοντά στους πολίτες, που αντιλαμβάνονται καλύτερα την προβληματική και που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ε, κατοίκων ε, των ε, περιφερειών αυτών προς το καλύτερο. Είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για τις μεταφορές, είτε για οτιδήποτε. Βέβαια οι περιφέρειες είναι αλήθεια ότι έχουν περιορισμούς κονδυλίων συγχρηματοδότησης κτλ. Συμφωνώ μαζί σας για το ρόλο των πόλεων, ότι είναι δηλαδή πολύ σημαντικός. Και είμαι ευγνώμων προς την Ολλανδική Προεδρία για τη σημασία που δίνει στο θεματολόγιο για τις πόλεις. Πράγματι, οι ευρωπαϊκές πόλεις, είτε πρόκειται για πρωτεύουσες, είτε πρόκειται για πιο μικρές πόλεις, 70% των ε, πολιτών μας ζουν στις πόλεις. Πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ευχαριστώ επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στηρίζει την εταιρική σχέση στην οποία και εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Φανίστεροι, για το ότι χρειάζεται δημόσια διαβούλευση για να δούμε πώς εφαρμόζεται η πολυδιάστατη διακυβέρνηση και εταιρική σχέση. Την επόμενη εβδομάδα θα συμμετάσχω στην Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Με ιδιαίτερη χαρά θα επανέλθω εδώ για να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι κάτι αναγκαίο. Υπάρχουν χώρες που έχουν την νοτροπία αυτή, τη συνήθεια αυτή τέτοιων προγραμμάτων και συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, τον ακαδημαϊκό χώρο, τα πανεπιστήμια κλπ. Αλλού, σε άλλες χώρες, ε, πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους πολίτες και η κεντρική δίκηση αποφασίζει μόνη της. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην συμμετοχή, την πραγματική συμμετοχή των τομικών και περιφερειακών αρχών στα επιχειρησιακά προγράμματα, κλπ. Ξέρετε ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο είναι εξάντε ε, υποχρέωση αυτή. Δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω μεμονωμένα σε όλες σας τις ερωτήσεις, αλλά θέλω να απαντήσω στον κύριο Γιάκοπτσιτς, ο οποίος ρώτησε κάτι που επανήλθε στη συζήτηση. Το ρώτησαν κι άλλοι. Θέλω λοιπόν να πω ότι κάθε χώρα μπορεί να οργανωθεί όπως επιθυμεί. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η οργάνωση αυτή και η εφαρμογή των προγραμμάτων να σέβεται τους κανόνες. Όταν πρόκειται για διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων υπάρχουν χώρες όπως η Πολωνία που είναι μια χώρα με κεντρική δίκηση που έχει καλές επιδόσεις στον τομέα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αλλά έχουμε και τη Γαλλία η οποία έχει περάσει σε ένα σύστημα αποκέντρωσης που επίσης λειτουργεί πολύ καλά. Συνεπώς κάθε χώρα μπορεί να οργανωθεί όπως το επιθυμεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η αρχή της εταιρική σχέσης από τις χώρες μέλη. Βάσει το άρθρου 5 των ε, ρυθμίσεων για το επενδυτικό ταμείο. Τώρα έρχομαι στο θέμα των ε, προσφύγων. Εμείς δεν υποχρεώνουμε καμία χώρα, καμία πόλη, καμία περιφέρεια να χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμείς την επιστολή αυτή τη στείλαμε σε όλους τους υπουργούς για να τους γνωστοποιήσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τον προγραμματισμό Ξέρουμε ότι εκπονήθηκαν πριν από ένα χρόνο τα προγράμματα. Η πρόκληση όμως η σημερινή που έχουμε το προσφυγικό δεν υπήρχε τότε. Η Ιταλία ήταν η μόνη χώρα η οποία ζήτησε λοιπόν την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ήδη έχουμε στείλει 220 εκατομμύρια ευρώ για να χτιστούν να φτιαχτούν κινητά νοσοκομεία, νηπιαγωγεία κλπ. Άλλες χώρες, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Γερμανία χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την ένταξη των ε, μεταναστών. Αλλά δεν υπάρχει καμία σύνδεση ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων και θεμάτων για τους πρόσφυγες. Άμεση τέτοια σύνδεση. Μία τελευταία διευκρίνηση τώρα. Με εκπλήσει που βλέπω ότι κάποιος από το UKIP λέει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι αναγκαία. Ξέρω ότι έρχεστε από μια λιγότερο αναπτυγμένη περιοχή, υποβαθμισμένη, η οποία υποφέρει επειδή κλείσανε ορυχεία εκεί. Ευχαρίστως να επισκεφτώ την περιφέρειά σας για να δείξουμε στους Βρετανούς πολίτες πώς συνεισφέρει η πολιτική συνοχής στην απασχόληση, στην κατάρτιση υπέρ της απασχόλησης και ότι υπάρχει αλληλεγγύη. Θέλουμε μια ενωμένη Ευρώπη. Ελπίζω η ιδέα αυτή να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση.